Uh, καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Άμυνας και Ασφάλειας. Η κυρία Φωτίγα μου ζήτησε να την αντικαταστήσω για αυτή τη συνεδρίαση λόγω υποχρεώσεων που έχει στην ε, εκλογική της περιφέρεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ε, διαδικασία. Έχουμε καταρχήν την έγκριση της τη διάταξης. Έχετε κάποια σχόλια σε σχέση με την τη διάταξη. Εγκρίνεται. Υπάρχει η ανακοινώση για την ε, διερμηνία που υπάρχει και Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Τα πρακτικά της 16 Μαρτίου και 20-21 Απριλίου. Έχετε σχόλια και αυτά τα εγκρίνουμε. Ναι, συγγνώμη. Περνάμε λοιπόν στο κύριο θέμα. Θέλω να καλωσορίσω τον υπονάβαρχο Βάλτε Μαρτιλιούσκο, ο οποίος είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης μαζί του είναι ο Τζονίζη Λόρια, ο ταξίαρχος Τζονίζη Λόρια, ο οποίος είναι ο διευθυντής υπεύθυνος για την επιμελητία. Πολλές φορές η υποεπιτροπή μας έχει επικρίνει το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ε, CSDP σε ό,τι τη σκέπασε ό,τι αφορά την εκπαίδευση έχει εμποδιστεί από την έλλειψη εξοπλισμού και έτσι δεν μπορούμε να βοηθούμε τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται σε κρίση να επιλύουν τα προβλήματα αυτά μόνες τους. Γι' αυτό θέλησαμε να θέσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Το Κοινοβούλιο πάντα προσπαθεί να <clears throat> βοηθήσει και με τον προϋπολογισμό αλλά και με πιο απτούς όρους να βοηθήσει τις προσπάθειες της ΚΕΠΑ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στο Κοινοβούλιο. Λυπάμαι για την ε, παρουσία των συναδέλφων ή καλύτερα για τη μη παρουσία ε, συναδέλφων. Αλλά εγώ μόλις ήρθα από το αεροδρόμιο και πολλοί συνάδελφοι έχουν πρόβλημα να έρθουν γιατί είναι μπλοκαρισμένο το αεροδρόμιο. Εγώ χρειάστηκα σχεδόν, σχεδόν δύο ώρες να έρθω και κάποιοι συνάδελφοι ελπίζω ότι θα έρθουν τα επόμενα λεπτά. Η πρωτοβουλία για το Capacity Building for Security and Development, το CBSCD, γνωστό ως ε, εξόπλησε και εκπαίδευση. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει τελματώσει λόγω διαθεσμικών δυσκολιών για δύο βασικά θέματα, την κατάλληλη νομική βάση και πρέπει να μας απασχολήσει αυτό που μας έχει απασχολήσει για πολλά χρόνια και επίσης το θέμα, όπως πάντα, της χρηματοδότησης. Το να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτά τα <clears throat> δύσκολα και ακαθόδη θέματα και να καταλήξουμε σε μια νομοθετική πρόταση για το CBS, CBSD. Υπάρχει ο μηχανισμός του Clearing House, ο μηχανισμός ε, κατά κάποιο τρόπο συμψηφισμού, ο οποίος φαίνεται ότι μας δίνει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για τον συντονισμό του στρατιωτικού υλικού, του εξοπλισμού, των υπηρεσιών, των μεταφορών και των άλλων στρατιωτικών στοιχείων και ικανοτήτων, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτό. Και στις 8 Φεβρουαρίου το, το Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε σε μια γενική αντιμετώπιση για το clearing house mechanism, και θα μας ενδιαφέρει πολύ να μάθουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό και σας ζητώ και πάλι την, την κατανόησή σας για την ε, ίσχυνη μας παρουσία. Νομίζω όμως ότι θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι. Χαίρομαι που είσαστε εδώ και μπορείτε να μας παρουσιάσετε αυτό το θέμα για το CHM, το Clearing House Mechanism και προφανώς μας ενδιαφέρει <clears throat> να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να ακούσουμε αυτά που έχετε να πείτε σε σχέση με το κατά πόσο αυτό ο σομιγαλισμό μπορεί να, να παράσχει μια λύση στα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει όχι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές και κύριε, και κύριοι, σε 10 λεπτά θα σας ενημερώσω όσον αφορά αυτή την σύλληψη που αφορά το Cleaning House που ε, στρατιωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, συλλαβή, ε, ξεκίνησω πρώτα από το ιστορικό πλαίσιο όσον αφορά την ιδέα που οδηγεί σε αυτόν τον μηχανισμό clearing house και να σας πω και τα αρχικά αποτελέσματα και κατόπιν να συνεχίσουμε στην ε, ουσία αυτής της σύλληψη και αυτής της έννοιας για την συνέχεια της παρουσίασής μας. Οπότε και εγώ θα σας ε, απαντήσω στις ερωτήσεις ακριβώς όπως και ο Σύρους που παρίσταται και επί τη βάση των όσων κάναμε που στήριζονται στην εμπειρία μας. Τον Ιούνιο του 2013 η στρατιωτική πρέπει να βρει ένα μηχανισμό τόσο ώστε να βοηθηθεί ο συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη, όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας με τη Δυτική Αφρική και επίσης την αφίσμα, δηλαδή κάποιες δυνάμεις που είχαν αναλάβει δράση στο Μάλι, στο οποίο το σοβούσε μια κρίση και επαφή με τις τοπικές ενόπλες δυνάμεις. Οπότε η εμπειρία μας από αυτές τις δραστηριότητε μας δείξε στο να κάτσουμε και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε παρόμοιες καταστάσεις. Δηλαδή κάτι το οποίο να είναι κατεπήγον, κάτι που να επιβάλλει συντονισμό και κάτι ε, το οποίο να είναι κατανοητό από όσους ε, εμπελέκονται στη σχετική επιχείρηση. Θα έπρεπε να υπάρξει επομένως μια συνεκτική απόκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό συζητείται επί αρκετού τσικοκαιρό. Αρχάς του 2015 ε, η Διεύθυνση για την Επιμελητία ασχολήθηκε με το θέμα και ε, είπαμε ότι θα πρέπει πρώτα-πρώτα θα πρέπει να καλυφθεί η προπόθεση του κατεπίδοντος από τους εταίρους μας και να υπάρχει συντονισμός ε, σε σχέση με τους πιθανούς δωρετές. Να αξιοποιήσουμε το στρατιωτικό προσωπικό όσον αφορά την εμπειρία, τις δυνατότητές του και κάτι επίσης άλλο από πλευράς οργανωτικής. Να λύσουμε το πρόβλημα του μόνιμου ημί διορισμού του προσωπικού που θα στελέχουν αυτή την επιχείρηση. Οπότε αυτά είπαμε ότι θα ε, ενεργοποιούνται όποτε χρειάζεται. Τέλος, όπως είπε και ο Πρόεδρος, εγκρίθηκε αυτή η υπόθεση το Φεβρουάριο του 2016. Τώρα, ξαναγυρίζουμε στο ιστορικό πλαίσιο. Το Clearing House ξεκίνησε 21 πρώτα του 2013 και είχαμε 19 αιτήματα και 14 ε, προσφορές για όπλα, πυρομαχικά, οχήματα, ε, εξοπλισμό ε, φυσικών προσώπων, κάτι το οποίο τον έλαβαν τα κράτη-μέλη, τα οποία εδόρισαν τα σχετικά και τα οποία πήγανε προς ΕΚΟΑΣ, αφήσμενοι προς τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλή και προς την αποστολή μας τέλος πάντων στη χώρα. Τα πρώτα πήγαν καλά, αλλά βέβαια κάποια αιτήματα δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Είχαμε σχετική προσφορά που μετά απεσήρθε και επίσης υπήρχε χρηματοδότηση από διαφορετικούς διάβλους με διαφορετικούς τρόπους. Και όσον αφορά τις πρώτες προσφορές προς το Clearing House, είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά τις επιχειρήσεις ε, ε μετακομιδής κλπ. Οπότε είπαμε να υπάρχει ένα κέντρο συντονισμού όσον αφορά κάποιο στρατηγείο για ε, ενέργειες μεταφορές στρατιωτικού χαρακτήρα. Το Clean House στήριξε την αφήση με την ECOAS και της ε, δύναμης του Μαλή ήταν μια εμπειρία θετική. Έδωσε στην Ένωση μια ιδέα του πώς είναι δυνατόν να υπάρξει συντονισμός της υποστήριξης από τους δωρητές. Δεν υπήρξαν ήδη πόροι, δεν υπήρξε ίδιος προϋπολογισμός σε σχέση με τον εξοπλισμό. Οπότε και όλα εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη και από τους άλλους εμπλεκομένους όσους θέλουν να στηρίξουν αυτή την υπόθεση. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ε, ένα τμήμα του υλικού το οποίο δόθηκε, δωρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Cleaning House. Τώρα, αυτό το οποίο γίνεται είναι να εξηγηθεί το πώς λειτουργεί το Cleaning House, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις της ΚΕΠΑ ή άλλου είδους εξωτερικές δράσεις. Διαδικασίες, λειτουργίες, όλα αυτά επιστρατεύονται όποτε ληφθεί η απόφαση ενεργοποίησης του κανονισμού. Οπουδήποτε τέλο πάντων ληφθεί η απόφαση συνεργοποίησης. Πάντως, ενεργοποιησης παντως παντα το κλίνιχα όσο αφορά κάποιες κατεπίγουσες περιπτώσεις. Ξεκινάμε τις ε, δωρεές, χρειάζεται συντονισμός και επιδιώκεται η αποφυγή επικαλύψεων για υλικό, για παροχή υπηρεσιών, για ε, μεταφορές ε, όσον αφορά τον εξοπλισμό και γενικά τις δυνατότητες των στρατιωτικών της Ένωσης. Οπότε το Clean House μπορεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει το υλικό που χρειάζεται για να υποστηρίξει εταίρους, να υποστηρίξει συνεργαζόμενες οργανώσεις, ό,τι χρειάζεται με έναν τρόπο αποτελεσματικό και συντονισμένο. Το Clean House είναι ανοιχτό σε όλους τους ενδυνάμει δωρητές και του ιδιωτικού τομέα, αν χρειάζεται, και ε, πρόκειται για τα κρατή-μέλη, πρόκειται για την ε, ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, την Επιτροπή, τριτά κράτη, διεθνεί οργανισμού όπω τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΝΑΤΟ. Και επίση έχουμε και κάποιου οργανισμού κυβερνητικού και μη κυβερνητικού. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το μηχανισμό πρόκειται να ετούνται αυτό το οποίο θέλουν σύμφωνα με τις αρχές του clearing house. Οπότε και ε, το cleaning House πρόκειται να είναι το μοναδικό σημείο επαφής και η ομάδα, η υπηρεσία του cleaning House πρόκειται να συμμετάσχει να δώσει οδηγίες, να καθοριστούν οι προτεραιότητες και έτσι να λειτουργήσει ο μηχανισμός του cleaning House και να είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής και συνεχώς να αναφερόμεθα σε όλους όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή. Οι δωρητές πολλές φορές το κάνουν αυτό ε, εκούσια και υπάρχουν και κάποια θέματα διοικητικά όπως εισαγωγή, αδειοδότηση εισαγωγών, αποθήκευση ε, και άλλα. The command Τώρα όσον αφορά τον κοινό έλεγχο και την σχετική απόφαση για αυτούς τους ελέγχους στα πλαίσια της ΥΠΑ της εκπροσώπου παρέχονται οι συμβουλές από τους στρατικούς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την, τι κατεύθυνση θα πάρουν οι δράση, τι θα γίνει και ο Γενικός Διευθυντής επίσης ε, συμβουλεύει και ενημερώνει τα κράτη-μέλη μέσω της ε, Στρατιωτικής Επιτροπής. Δεν χρειάζονται παραπάνω πόροι προς τούτο. Όσο αφορά το προσωπικό, όσο αφορά τους πόρους, χρησιμοποιούνται οι πόροι οι οποίοι ήδη διατίθενται για το στρατιωτικό προσωπικό της Ένωσης και βέβαια όλα εξαρτώνται από την ε, σχετική δραστηριότητα. Εάν καλύπτεται εντάξει, αν όχι ε, επιδιώκεται η κάλυψή της και υποστήριξή της τώρα. Εδώ έχουμε το πώς ε, συγκροτηθεί αυτός ο μηχανισμός σε σχέση με το αποδέκτη και τώρα θέλουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η δουλειά από την υπατή εκπρόσωπο όσον αφορά αυτή την μονάδα και το στρατηγικό προσωπικό δεν εμπλέκεται στην ε, εκτέλεση των ε, δωρεών. Εμείς έχουμε ρόλο συντονιστικό για τον μηχανισμό. Εξαρτάται τι δορίζεται, ποιος είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας και συνοψίζοντας δεν είναι η λύση του προβλήματος το κλινικά είναι μέρος της λύσης. Βεβαίως και η υπόθεση αυτή επιδέχεται βελτίωση. Θα πρέπει τα κρατημέλη να, δωρε, να δωρήσουν, αλλά θα πρέπει και να βοηθήσουν γενικότερα. Σας ευχαριστώ και ευχαρίστω να απαντήσω τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους για τυχόν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και έχω κάποια ερωτήματα. Αυτό το σύστημα, αυτός ο μηχανισμός στηρίζεται στις συνεισφορές των ε, κρατών μελών. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτές τις ε, συνεισφορές και θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ε, δυνατότητα να συνεισφέρει και πόσο σε εξοπλισμό κτλ. Έπειτα, όσον αφορά την την επίλυση κρίσεων. Ε, τι έχετε να πείτε για τις ανάγκες που προκύπτουν. Και τι συμβαίνει με τον ε, προϋπολογισμό. Εδώ στο Κοινοβούλιο ε, ένα από τα ερωτήματα που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό. και το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους ε, πόρους για θέματα ασφάλειας. Και οι πόροι αυτοί, εάν θα πρέπει να είναι ξεχωριστοί ή Ευρωπαϊκή; Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω στην ερώτηση του συναδέλφου. Υπονάβαρχε, ε, μας μιλήσατε για τον μηχανισμό αυτό, όμως ε, έχουν παρατηρηθεί κάποια προβλήματα σε αυτόν τον μηχανισμό. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιήθηκε στο Μάλι. Τώρα, οι εμπειρίες σε σχέση με την χρήση του μηχανισμού αυτού στην περίπτωση του Μάλι, τι σας έχουν διδάξει. I don't know which... Δεν ξέρω ποια γλώσσα να χρησιμοποιήσω για να σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω στα αγγλικά λοιπόν, αν δεν σας πειράζει. Κύριε Ζέμκα, να απαντήσω στη δική σας ερώτηση πρώτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε σε επιχειρήσεις στην Αφρική. Κατά κύριο λόγο, όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή βρίσκονται να εξελίξει έξι τέτοιες επιχειρήσεις και υπάρχει κάποιος διακανονισμός σε σχέση με την χρήση του μηχανισμού ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε εστιάσει στην στρατιωτική πτυχή, θα μπορούσαμε όμως να επεκτείνουμε τον μηχανισμό. Ελπίζουμε να επεκταθεί ο μηχανισμός αυτός και σε μη στρατιωτικού τύπου επιχειρήσεις. Το πρόβλημα που εντοπίσαμε, αρχίζοντας από την περίπτωση του Μάλι, ήταν ότι αρχικά το σχέδιο ήταν να αναπτύξουμε μία ε, αποστολή κατάρτισης στο Μαλί. Υπήρχε μία αφρικανική αποστολή ήδη Και το πρόβλημα που συναντήσαμε ήταν ότι υπήρχε μεν η γνώση, αλλά όχι ο εξοπλισμός. Είχαμε λήψει εκεί. Και εστιάσαμε λοιπόν στην στήριξη των ε, άλλων φορέων για εξοπλισμό. Τώρα, αν τα κράτη-μέλη μας ε, προσέφεραν εξοπλισμό, υπήρχε και ένα πρόσθετο πρόβλημα του πώς αυτός θα μεταφερθεί. Στην περίπτωση του Μάλι, όπως σας είπα, υπήρξαν 19 αιτήματα και 14 προσφορές από τα κράτη-μέλη. Και όσον αφορά τα συγκεκριμένα νούμερα, ίσως εσείς και οι συνάδελφοι να μπορούσατε να απαντήσετε καλύτερα. Η πλειοψηφία, αν όχι όλοι, όλες οι προσφορές, εν τέλει μεταφέρθηκαν στην αποστολή στο Μαλί και έπειτα στις ίδιες τις ένοπλες δυνάμεις του Μαλί. Μπορούμε δηλαδή να πούμε πως ε, δεν ήταν απόλυτη επιτυχία, όμως υπήρξε επιτυχία ως ένα σημείο. Τώρα, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και την ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στις χώρες στις οποίες είχαμε αναπτύξει αποστολές. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να μεταφερθεί γνώση, αλλά να μεταφερθούν και δυνατότητες. Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εξοπλισμός. Και όπως ε, προανέφερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ίδιους πόρους για αυτό και σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τον μηχανισμό Αθηνά, ε, ο οποίος αφορά το κόστος μιας στρατιωτικής, ε, στρατιωτικής επιχείρησης. Και στην περίπτωση αυτή δεν αφορά τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Γι' αυτό λοιπόν εξαρτώμαστε από την γενοδορία των κρατών μελών. Και στην περίπτωση του Μάλι ζητήσαμε βοήθεια και είχαμε μερική επιτυχία. Τώρα, σχετικά με την προθυμία των κρατών μελών να στηρίξουν αυτή την πρόταση, μπορώ να πω ότι στην περίπτωση του Μάλι καταφέραμε να διαχειριστούμε μόνοι μας την ε, κρίση αυτή. Είχαμε εμπειρογνωμοσύνη, είχαμε γνώση, είχαμε το ανθρώπινο δυναμικό για να το πράξουμε. Όμως για το μέλλον δεν είχαμε ακόμα την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες του μηχανισμού. Όπως σας είπα, είναι κάτι που έχει εγκριθεί πρόσφατα και εφαρμόστηκε μόνο μία φορά στο Μάλι. Τέλος. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Μα γι' αυτό σας έκανα λόγο για την ανάπτυξη ικανοτήτων, για την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Και αυτή η ιδέα για μια κοινή ε, επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών υπήρχε από πολύ καιρό. Προσπαθούσαμε όμως να βρούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτήν την πρόταση. Προς το παρόν δεν κάνουμε λόγο ε, για, εξοπλ, για στρατιωτικό εξοπλισμό, όπλα, πολεμικά, οπλικά ε, συστήματα. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσω του μηχανισμού Αθηνά για τα απλά ζητήματα, δηλαδή καρέκλες, τραπέζια, τέτοιου είδους εξοπλισμός ε, για αποστολές κατάρτισης, εκπαίδευσης. Υπάρχει πρόβλημα με τις στολές για τους στρατιωτικούς, δεν επαρκούν. Βασικά πράγματα δηλαδή. Πού αλλού αντιμετωπίσαμε προβλήματα, στις υποδομές μιας τέτοιας επιχείρησης ε, κατάρτισης. Και δεν ε, μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες ε, μέσω του μηχανισμού Αθηνά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποια λύση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Γι' αυτό λοιπόν από αυτή την οπτική γωνία Σίγουρα μπορώ να πω ότι πρέπει να βρούμε μια πηγή χρηματοδότησης. Τώρα, ε, για να απαντήσω στη δική σας ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, η αφετηρία ήταν το μαλλί. Και πράττουμε βασιζόμενοι στις εμπειρίες που αντλήσαμε από εκεί. Σίγουρα αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα στη Σομαλία, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και υπάρχει ανάγκη εξοπλισμού, ο οποίος θα μπορέσει να στηρίξει τις διάφορες αποστολές μας, αποστολές ε, εκπαίδευσης σε αυτές τις χώρες, της μη στρατιωτικού τύπου. Γι' αυτό λοιπόν μπορώ να σας αναφέρω μόνο την περίπτωση του Μάλι. Γιατί είναι βασισμένη σε γεγονότα και να την μεταφέρω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πιο θεωρητικό για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Με λίγα λόγια, είναι ένας απλός μηχανισμός ο οποίος είχε αποτέλεσμα όταν εφαρμόστηκε και εμείς μπορούμε να δούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε, ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο στο μέλλον. Δεν είναι θέμα δηλαδή πόρων, χρημάτων, είναι θέμα γνώσης, εμπειρογνωμοσύνης και της ικανότητας να συνδέσουμε διάφορες πηγές. Τώρα, όσον αφορά την εφοδιαστική, τη μεταφορά, είναι και αυτοί οι παράγοντες πάρα πολύ σημαντικοί. Διότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες ήταν πρόθυμες να προσφέρουν εξοπλισμό ή, δια, ή άλλου τύπου δωρές, όμως ήταν δύσκολο αυτό να μεταφερθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή έχουμε και τον ταξίαρχο <clears throat> Ρίτζι, ίσως θέλετε να προσθέσετε κάτι. Διακεκριμένα μέλη του Κοινοβουλίου, καλό απόγευμα. Για να συμπληρώσω αυτό που είπε ο υπονάβαχος Κουσκό για την εμπειρία μας στο μαλή. Ο στόχος του Clearing House ήταν διπλός. Πρώτα απ' όλα να διευκολύνουμε την ταχεία ανάπτυξη <clears throat> της αποστολής με ηγεσία της Αφρικανικής Ένωσης και δεύτερον να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εκπαιδευτική αποστολή στο Μαλί. <clears throat> Μετά από ένα αρχικό διάστημα που ήταν απαραίτητο για την οργάνωση, τη δημιουργία των διαδικασιών του Clearing House. Το επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την <clears throat> Στρατιωτική Επιτροπή για να εγκρίνει αυτή την αποστολή. Είχαμε μια θετική απάντηση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχαν 55 C17, τα οποία είναι 50 μάλλον C17 που είναι αεροπλάνα αερομεταφορών Μεγάλη χωρητικότητας από τη Σουηδία. Μετά άρχισαν να κουράζονται οι δωρητές. Επεκράτησε λεγόμενη κόπωση των χορηγών και γι' αυτό μία από τις βασικές ε, ε, προσπάθειες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να δώσουμε στους εκπαιδευόμενους τουλάχιστον <clears throat> τέντες για τη στέγασή τους, μπότες, στολές και όλα αυτά με την εργοποίηση του μηχανισμού Αθηνά. Επομένως, όπως είπε και ο, ο μπορεί το μηχανισμός του Clearing House να αντιμετωπίσει πολύ συγκεκριμένες ενέργειες. Αλλά η δημιουργία ικανοτήτων είναι κάτι το ευρύτερο, χρειάζεται, <clears throat> όπως είναι και στο Μαλί, να ξαναφτιάξετε τις ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά από το μηδέν. Είχαν διαλυθεί μετά από το πραξικόπημα στο Μαλί οι ένοπλες δυνάμεις είναι απαραίτητο λοιπόν να αντιμετωπίσει κανείς το θέμα ηγεσία και δημιουργία ιεραρχία και χρειαζόνται τα πάντα σε μια τέτοια περίπτωση. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου για τον εξοπλισμό, καταγραφής και ελέγχου του εξοπλισμού, συντήρησης του εξοπλισμού και εξασφάλιση μιας βιώσιμης ικανότητας η οποία μπορεί να επιτευχθεί από τις ενόπλες δυνάμεις του Μαλή και αυτό γίνεται πάντα σε μια εταιρική σχέση. Αλλά αλλιώς κινδυνεύουμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι δημιουργούμε μια κατάσταση εξάρτησης όπου οι άλλοι μας βλέπουν μονάχα σαν πηγή ελεημοσύνης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει και η συμμετοχή των ε, αποδεκτών και των δικαιούχων σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Και πάλι. Και απολογούμε που μπαίνω και πάλι σε αυτό το θέμα σε πιο πολύ λεπτομέρεια. Εγώ πήγα στο Μαλί για να δω αυτή την ε, επιχείρηση εκπαίδευσης. Βέβαια, άμα θέλει κανείς να βοηθήσει και βλέπει μετά ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, αυτό είναι κάτι το συντριπτικό. Αναρωτιέμαι κατά πόσο άλλαξε η κατάσταση με αυτή την αποστολή. Δεν μιλάμε για εξοπλισμό, για όπλα και τέτοια πράγματα. Και αυτή είναι μια περιοχή του κόσμου αυτοί οι οποίοι έχουν τον έλεγχο των όπλων, πολλές φορές δεν ήταν καν στρατιωτική. Ήταν καταστροφική κατάσταση. Αλλά το ερώτημά μου είναι σε ποιο βαθμό αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος γίνεται βέβαια σε περιστασιακό επίπεδο, αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο όπου εσείς έχετε συλλέξει μία σειρά από στοιχεία τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν. Ποια είναι η κατάσταση τώρα με αυτή την αποστολή. Σε ποιο βαθμό είναι μια λειτουργούσα επιχείρηση που βασίζεται σε επαρκή επίπεδα υποδομών για να μπορέσει να αναπτύξει μια νέα δομή για, το, για τη σπονδυλική στήλη του στρατού στο Μάλι με τη δημιουργία αξιωματικών παραγματος έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με αυτά που συνέβησαν πέρσι ή απλώς ρίχνουμε μία σταγόνα στον ωκεανό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εάν μπορώ. Η ασφαλευσικά είναι ένα προαπαιτούμενο για να μπορέσει να προχωρήσει οποιαδήποτε ενέργεια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια πρωτού περάσουμε στο επόμενο επίπεδο για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία ικανοτήτων. Ο μηχανισμός του Clearing House εισήχθη στην αρχή της ε, αποστολής μας στο Μαλί στην αρχή βοήθησε. Τώρα, δεν ε, χρησιμοποίησαμε αυτό το μηχανισμό πλήρως, γιατί δεν υπήρχαν προσφορές από τα κράτη-μέλη για να μας δώσουν εξοπλισμό ή τεχνογνωσία ή οποιοδήποτε το οποίο θα μπορούσε να δοθεί Προ το στατό και την αεροπορία του Μαλή. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και όπω είπα προηγουμένω. ήταν πραγματικά οδυνηρή η κατάσταση στο Μαλή. Εμείς τονίζουμε πάντα ότι οποιαδήποτε προσφορά, οποιαδήποτε δωρεά μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση, γιατί στο Μαλή τα πράγματα δεν είναι όλα αρνητικά. Το στρατόπεδο εκπαίδευση του Κοντικόρο είναι καλά εξοπλισμένο και προς το παρόν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την αποστολή εκπαίδευσης και να χρησιμοποιήσουμε όλη την ικανότητα που έχουμε για να εκπαιδεύουμε τους, ε, στρατιωτικ... τους στρατιώτες και στρατιωτικούς κοντά στους στρατώνες τους. Αλλά στη Σομαλία τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί εκεί οι συνθήκες εκπαίδευσης στους καταβλισμούς είναι πάρα πολύ ανεπαρκείς. παρά τα χρήματα τα οποία δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και φυσικά αρμόδια για τη δημιουργία και την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων, και που είναι αρμόδια για την καλή κατάστασή τους και την πληρωμή των στρατιωτών ή των εκπαιδευομένων, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα σε πιο καθημερινή βάση. Υπάρχει η ανάγκη λοιπόν να υπάρξει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο πιο οργανωμένο τρόπο το clearing house, ο μηχανισμός του clearing house είναι για έκτατη, για κατεπίγουσα αντιμετώπιση. Όταν πρόκειται για από πιο καθημερινά θέματα τα οποία χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται οι πιο κλασικές και συμβατικές λύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Για την Επιτροπή μας αυτό θα είναι θέμα που θα μας απασχολήσει μονίμως. Και θεωρούμε και εμείς και το Κοινοβούλιο ότι αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκού κύρους. Ε, είναι θέμα το οποίο αναβρώνει ή όχι την εικόνα μας στην Αφρική και αλλού. Άρα θα πρέπει η Επιτροπή μας να φροντίσει παγίως να συζητάτε αυτό το θέμα γιατί όπως έχουμε και το πολιτικό σκέλος θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει και από πλευράς μια ρύθμιση γιατί άλλωστε από πλευρά τα πράγματα σχετίζονται με πιο μεγάλη ανάληψη κινδύνου, είναι πιο κατεπήγοντα. Είναι δηλαδή μια κατάσταση, μια ρύθμιση που θα υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Ευχαριστούμε πολύ ε, κύριε Ναύαρχε, κύριε Ταξιάρχε. Σα ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι ε, είστε πιστοί στο καθήκον σας ε, σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και ότι δεν έχετε και τόσο μεγάλη υποστήριξη ε, από πλευράς υποδομής, από πλευράς πόρων. Και πάλι σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Thank Κυρίες και κύριοι, μετά το μικρό διάλειμμα να δούμε στις 4.30 το επόμενο θέμα της μεσής διατάξεως. Θα έχουμε την Επιτροπή για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα ασφάλειας και άμυνας για τη σχετική πρόταση δηλαδή. Όμως θα κάνουμε διάλειμμα μια που για τότε έχει προγραμματιστεί να γίνει η προσέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα σε περίπου τρία τεταρτάκια.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 So, Κυρίες και κύριοι, σχεδόν 4.30 και πιστεύω πως πρέπει να συνεχίσουμε με το δεύτερο σημείο της ημερησίας διάταξης, προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της ΚΕΠΑ. Έχουμε εδώ τον Έλενα Λέξη, προϊστάμενο τη διοικητική μονάδα για άμυνα αεροδιαστημική και ναυτιλία από τη ΔΕΛΤΑ Grow. Πιστεύω ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι, ένα, είναι από τα βασικότερα προγράμματα τα οποία ε, αφορούν το Κοινοβούλιο όχι μόνο για θέματα άμυνας αλλά και για θέματα έρευνας. Και χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που έχουμε σήμερα ανάμεσά μας τον ε, πατέρα αυτής της ιδέας, τον κύριο Γκάλερ, Είναι ένας λοιπόν από τους πατέρες αυτής της ιδέας. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ ως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια σημαντική φιγούρα πίσω από την πρόταση αυτή. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν θα ήθελα να σας δώσω το λόγο έτσι ώστε να μας παρουσιάσετε μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. με την πρόταση που πρόκειται να δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν κάνω λάθος, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις. Το Συμβούλιο Γερμανία-Γαλλία τουλάχιστον σίγουρα. Και έχετε αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε Τα θέματα της ε, άμυνας αποκτούν μια, μια σημασία όλο επαυξανόμενη και φυσικά θα μας απασχολήσουν και ως το τέλος του χρόνου. Έχουμε ενεξελίξει πολλά έγγραφα το οποία είναι πολύ σημαντικά όπως είναι η στρατηγική της κυρίας Μογκερίνη για να παρουσιαστεί προς το τέλος Ιουνίου η Λευκή Βίβλος η οποία είναι συνέχεια για τη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων, το σχέδιο δράσης κομισιών, σε ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα για το δεύτερο εξάμεινο του 2016 και την προπαρασκευαστική δράση η οποία είναι περισσότερο προθυμένη. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουν υπάρξει ήδη στο παρελθόν πολλές πρωτοβουλίες για τα θέματα αυτά. Η τελευταία ήταν η ανακοίνωση της Κομισιόν το 2013 αν δούμε την κατάσταση λοιπόν αυτή, τι έχει αλλάξει από σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία, αν σκεφτούμε το διεθνές πλαίσιο, το οποίο δυστυχώς δεν έχει φεφ βελτιωθεί και απαιτεί απαντήσεις από εμά. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και δεύτερον, η Ευρώπη θέλει να δώσει χρηματοδότηση περισσότερη για την αμυντική έρευνα. Πάρα πολύ σημαντικό γιατί παραδοσιακά δεν υπήρξε κοινωτική χρηματοδότηση για τα ερευνητικά θέματα στον τομέα της καθαρής άμυνας. Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή και επομένω αυτή η προπαρασκευαστική δράση είναι πολύ σημαντική αυτή κάθε αυτή και για την συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί μετά από αυτήν. Όταν λέμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο. Νομίζω ότι είναι σαφές και το καδεκνή και η έκθεση της ομάδας προσωπικότητων που δημιούργησε η κυρία Μπιενκόφσκα που έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σαν στόχο να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την έρευνα και δεν θα πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ της ε, εθνικής Έρευνα και τη ενωσιακή έρευνα Θα πρέπει να είναι συμπληρωματικέ οι δύο αυτέ ενέργειε. Όπω είπε η ομάδα των προσωπικότητων, θα πρέπει να υπάρχει μια σημαντική προσθέμενη αξία από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι αφορά την έρευνα. Οι προσωπικότητε επίση τόνισαν σε μεγάλο βαθμό το γεγονό ότι πρέπει να υπάρξει και μια σύνδεση μεταξύ τη έρευνα, Αφενό, και τη ανάπτυξη αφετέρου. Ο στόχος δεν είναι μοναχα η έρευνα, αλλά μία αλυσίδα που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και θα επιτρέψει να καταλήξουμε σε ένα προϊόν που τελικά μπορούν να αγοράσουν το κατημέρι και να χρησιμοποιήσει ο στρατός. δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε έρευνα η οποία δεν οδηγεί σε αυτά αποτελέσματα. Κύρια θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στα πλαίσια αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης και σε ό,τι αφορά το επίπεδο προβληματισμού μας. Ένα βασικό στοιχείο είναι η διακυβέρνηση η οποία πρέπει να δημιουργηθεί για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Η Κομισιόν βασίζεται στους ε, παραδοσιακούς μηχανισμούς με κάποιες τροποποιήσεις. Γι' αυτό δημιουργήσαμε μια επιτροπή προγράμματος η οποία δεν είναι ακριβώς κλασική επιτροπή προγράμματος αλλά η οποία συναθρίζει τα κράτη-μέλη, κάτι που είναι σημαντικό γιατί έτσι έχουμε και την άποψη των κρατών μελών. Επιπλέον συμμετέχουν σε αυτήν ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Φορέας, ΕΝΤΑ, που δίνει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για να ενισχύσει τις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή θεσπίστηκε το Δεκέμβριο του 2015. Έχουν λάβει χώρα οι δύο σημαίνες συνεδριάσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν και στο 2016. Δεύτερη σημαντική ομάδα είναι η συμβουλευτική ομάδα, όπου είναι οι εμπειρογνώμονες του τομέα και θα δημιουργηθεί στις επόμενες εβδομάδες. Εμείς ε, περατώνουμε τον κατάλογο των μελών αυτής της συμβουλευτικής ομάδας με στόχο να συγκεντρώσουμε άτομα με ιδιαίτερες ε, δεξιότητες από τον πανεπιστημιακό χώρο, εμπειρογνώμονες, από την βιομηχανία, που θα προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους για το θέμα αυτό. Εάν θέλουμε αυτή η δράση να είναι επιτυχής, τότε θα πρέπει κάπως να την αποδεχτεί και η βιομηχανία και να την εγκολποθεί. Θέλουμε λοιπόν να είναι παρούσα η βιομηχανία και να μας δώσει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για να προχωρήσει αυτή η προπαρασκευαστική δράση. Έχουμε δημιουργήσει επίσης, όπως είπα, μια στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Φορέα, με τον οποίο έχουμε σχεδόν καθημερινά συναντήσεις. Ο φορέας αυτός έχει μια τεχνική τεχνογνωσία που η Κομισιόν δεν έχει. Είναι απαραίτητη λοιπόν η συνεργασία στον τομέα αυτό για να μπορέσουμε να φέρουμε σε αίσιον πέρα σε αυτό το εγχείρημα. Η συνεργασία αυτή έχει ενισχυθεί περαιτέρω και με το πιλωτικό σχέδιο που ξεκίνησε στο τέλος του 2015 Έχουμε μια <clears throat> συμφωνία ήδη με τον φορέα ε, για τα αμυντικά θέματα για το πιλωτικό σχέδιο. Το πιλωτικό αυτό σχέδιο έχει περιορισμένη χρηματοδότηση από τον προπολογισμό, αλλά μόλον τούτο το σχέδιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι επιτρέπει να δημιουργηθεί μια δομή και μια μορφή συνεργασίας με τον φορέα άμυνας, με τον ΕΝΤΑ, επιτρέπει να δοκιμάσουμε μια σειρά από παρεμβάσεις να αντιμετωπίσουμε θέματα παραγωγικά πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πιλωτική αυτή ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική, έχει προχωρήσει ήδη. Συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής ε, σχεδίων και ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει προβλεφθεί. Για τις συγκεκριμένες μορφές που θα πάρει αυτή η προπαρασκευαστική δράση, φυσικά θα είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται να ανοίξει και σε τρίτες χώρες αυτή η συνεργασία. Ίσως θα υπάρξει μία εξαίρεση για την Ορβηγία, η οποία είναι πολύ κοντά στα κρατημέλη σε θέματα άμυνας. Μπορούμε λοιπόν να διευρύνουμε αυτή την ε, δράση και στην Ορβηγία. Μία άλλη σημαντική πτυχή είναι η πτυχή των πνευματικών δικαιωμάτων που θα προκαθορίσει και την επιτυχία την αποτυχία της προπαρασκευαστικής δράσης και των ερευνητικών προγραμμάτων. Γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Για τα προγράμματα έρευνας, τα οποία θα διαχειριζόνται τα κράτη-μέλη, η κατάσταση είναι απλή. Γιατί στις περισσότερες φορές τα κράτη-μέλη οργανώνουν διαδικασίες προσφορών σε ανταγωνιστικό επίπεδο και τα κράτη-μέλη ουσιαστικά είναι οι εντολοδόχοι και οι αγοραστές της ε, έρευνας. Όταν το κάνουν αυτό είναι και οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε σχέση με αυτά τα πνευματικά δικαιώματα. Για την προπαρασκευαστική ενέργεια όμως το ερώτημα είναι, είναι αν θα έχουμε μονάχα χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις ή αν θα έχουμε ε, και περαιτέρω παρεμβάσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα. Μέσα στα πλαίσια του προβληματισμού με τα κράτη-μέλη, η τάση είναι γενικά να περιοριστεί η δράση αυτή σε ε, χορηγίες που είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν σε μια τέτοια προπαρασκευαστική δράση, δηλαδή η Κομισιόν να, να χρηματοδοτήσει την ε, έρευνα με καθαρές χορηγίες. Το επόμενο ερώτημα είναι όταν έχουν εφαρμοστεί αυτά τα προγράμματα, όταν τα πορισμάτια των ερευνών έχουν συλλεγεί, τι είδους περαιτέρω προγράμματα μπορούμε να έχουμε. Μας λένε τα κρατημέλη ότι αυτή η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί με χρήματα του δημόσιου τομέα, οπότε θα πρέπει και τα κρατημέλη να επωφεληθούν από αυτά τα πορίσματα της έρευνας για να συνεχίσουν με προγράμματα follow-up. Μας λένε οι επιχειρήσεις, ε όχι όμως, αυτή η έρευνα είναι δικιά μας. Εμείς έχουμε βέβαια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι μια επιδότηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι δικά μας και μόνο. Πώς θα εξασφαλίσουμε λοιπόν την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο αντιρρόπων θέσεων. Κατανοούμε την άποψη των επιχειρήσεων. Τα πνευματικά δικαιώματα, ιδίω στον τομέα τη ε, έρευνα είναι βασικό ενεργητικό στοιχείο μια επιχείρηση. Δεν μπορούμε να πούμε σε μια επιχείρηση να εγκαταλείψει τα δικαιώματά τη και να τα δώσει μονάχα στο δημόσιο τομέα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που είναι το γεγονό ότι αν εμεί χρηματοδοτούμε την έρευνα, περιμένουμε να υπάρξουν και θετικές απολύξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια για τα προγράμματα έρευνας. Ούτως ή άλλως λοιπόν θα πρέπει τα αποτελέσματα της έρευνας να χρησιμοποιηθούν για να υλοποιηθούν περαιτέρω προγράμματα που θα οδηγήσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Πού είναι η σωστή ισορροπία. Εκεί η ομάδα προσωπικότητων της κυρίας Βιενκόφσκα μας ε, παρέθεσε μία σειρά από επιλογές στην εκθεσή τους. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι επιλογές. Αλλά πρέπει ακόμα να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη που θα θέλανε πράγματι να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Για την Κομισιόν όμως η προστασία των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αν η προπαρασκευαστική δράση δεν ανταποκρίνεται βέβαια στις επιθυμίες των κρατών μελών κινδυνεύουμε να προσκρούσουμε σε μια αποτυχία που δεν είναι και ο στόχος μας. Μία άλλη σημαντική πτυχή είναι ο προπολογισμό. Που αφορά αυτή την προπαρασκευαστική ενέργεια, η δράση και οι επαφέ στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξελίσσονται και ελπίζουμε ε, σύντομα να έχουμε μια τοποθέτηση όσον αφορά πρόταση για τον προπολογισμό, αλλά βέβαια οι αρχέ του προϋπολογισμού θα πρέπει να αποφασίζουν σχετικώ είναι, είπαν, προπαρασκευαστική δράση, ενέργεια, πότε υπάρχουν περιορισμοί από τον ε, προπολογισμό. Βέβαια, πέραν αυτού θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια ε, όσον αφορά τον προπολογισμό, γιατί αξίζει, ε, κοστίζει πολύ η έρευνα όσον αφορά την άμυνα. Άρα θα πρέπει να δεσμευθούν πόροι σχετικώ. Και δεύτερον, από πολιτική πλευρά, εάν θέλουμε κάτι να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να στείλουμε θετικό μήνυμα. Και όσον αφορά το Υπουργείο Άμυνα και την βιομηχανία. Εάν θέλουμε από πλευρά κοινότητα κάτι να φτιάξουμε, θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη δημοσιονομική δέσμευση. Άρα θα πρέπει να γίνουν επαφές τόσο να φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές νούμερο. Τώρα όσον αφορά τα βασικά θέματα που θα καλύψει αυτή η προπαρασκευαστική δράση και επ' αυτού έχουμε τις προσωπικότητες που θα καλύψουν σημαντικούς τομείς, με κάποιον για επίδειξη γιατί νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο ρόλος, γιατί μιλάμε για μια μικρή περίοδο σχετικά. Μέσα σε τρία χρόνια θα πρέπει να επιδείξει και να αποδείξει την προσθεμένη αξία της Ευρώπης. Εάν ξεκινήσουμε λοιπόν την βασική έρευνα, τότε τι θα γίνει. Σε δέκα χρόνια τι θα έχουμε κάνει. Επομένως χρειάζεται κάποιος που να μπορέσει να αποδείξει το ζητούμενο από πλευρά τώρα ε, και κριτικής, από πλευράς λειτουργικότητα και αυτό είναι σημαντικό. Και εδώ έχουμε τα σχετικά στάνταρ και πρότυπα πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε από πλευράς τώρα διαδικασίας και χρονοδιαγράμματος εμείς αυτό το οποίο σχεδιάζουμε είναι να υπάρξει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου να γίνει η σύνθεση της ακολουθητέας ε, πορείας και μιλούμε για το δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους για αυτή την ανακοίνωση. Ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει το πότε. Μάλλον θα είναι κομμάτι του πακέτου με το πρόγραμμα δράσης και λοιπόν πρωτοβουλειών, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα για τα σαρχάς του 17. Αυτά όσον αφορά την προπαρασκευαστική δράση, Πρόεδρε. Ερώτηση. Κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλέξης για την παρουσίασή σας. Ως ε, μέλος αυτής της ομάδας λοιπόν προσωπικότητων θα ήθελα να σας ε, διαβεβαίωσω ότι εμείς στηρίζουμε απόλυτα αυτό το έργο για το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και ελπίζουμε να αρχίσουμε σύντομα με την έρευνα και την ανάπτυξη για θέματα άμυνας. Ε, φυσικά υπάρχουν και ερωτήματα όσον αφορά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ως προς τις προτάσεις που μας παρουσιάσετε για αυτά τα προπαρασκευαστικά μέτρα. Η κυρία Μπιενκόφσκα ήρθε πέρυσι τον Ιούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας μίλησε για θέματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και ο πρόεδρος Μπούζεκ αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα που ε, είχε αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πιλωτικά προγράμματα. Πριν από μερικές εβδομάδες όμως είδαμε ότι οι προθεσμίες άλλαξαν και ότι, δόθηκε, και ότι αναβλήθηκε ε, αυτή λοιπόν η παρουσίαση. Έχουν σημειωθεί λοιπόν καθυστερήσεις. Αυτές λοιπόν οι προπαρασκευαστικές δράσεις έχουν κάποιες ασάφειες ως προς το χρονοδιάγραμμα και θα ήθελα να μου πείτε πιο συγκεκριμένα πότε πρέπει να περιμένουμε τι. Μετά, στην αντίστοιχη έκθεση αναφέρεται η δημιουργία ενός ε, μια συμβουλευτική επιτροπή. Ε, τι γίνεται, που βρισκόμαστε με αυτή τη συμβουλευτική επιτροπή. Τώρα, από πέρυσι το Δεκέμβριο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει και μία υπο Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποιοι συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή, πόσες συνεδριάσεις έχουν γίνει, ποια είναι τα θέματα που συζητήθηκαν και εάν υπάρχουν αποτελέσματα, ποια είναι αυτά για αυτήν την Επιτροπή ΕΣΕΦ. Γνωρίζετε επίσης πως είναι έτοιμα και της Γαλλίας και της Γερμανίας να δημιουργηθεί ένα δίκτυο όπου θα ε, διατίθενται κονδύλια για τα επόμενα χρόνια. Πώς εσείς έχετε σκοπό να υλοποιήσετε ε, αυτή την πρόθεση. Και αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή, από ποιους θα αποτελείται, θα συμμετέχει η βιομηχανία και ο πανεπιστημιακός χώρος. Και όσον αφορά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν αυτές οι προπαρασκευαστικές δράσεις, αυτά θα οργανωθούν σε υποομάδες. Το Δεκέμβριο πέρυσι υπήρξε μια έκκληση προς τα κράτη-μέλη να διατυπώσουν τις επιθυμίες τους και τις δικές τους προτάσεις για αυτά ε, για αυτές τις ομάδες και να κάνουν προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα. Ε, όμως γιατί δεν απευθυνθήκατε άμεσα και απευθεία στα κράτη-μέλη για αυτά τα προγράμματα. Μετά, θα με ενδιαφέρε να μου πείτε αυτές οι προπαρασκευαστικές δράσεις πώς θα επιτύχουν την συγχρηματοδότηση από τα κρατημέλη. διότι μέσω της σύγχρηματοδότησης τα κράτη-μέλη έχουν την ε, δυνατότητα να ε, δεσμεύσουν κάποια κονδύλια που θα αφιερωθούν σε αυτά τα προγράμματα. Τι προβλέπετε λοιπόν για αυτό. Εμείς από τη δική μας πλευρά θα στηρίξουμε κάτι τέτοιο, αλλά περιμένω να μου απαντήσετε για τις, ε, με τις δικές σας ε, εκτιμήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσάνκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ιδιαίτερα μάλιστα, διότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, επιτέλους ήρθε η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει την έρευνα στον χώρο της άμυνας. Και γνωρίζουμε επίσης ότι υπήρξαν προβλήματα στη χρηματοδότηση στο παρελθόν. Δεν μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει αυτή την έρευνα. Όμως, τώρα, όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, καταλήξει στο να συμμετέχουν οικονομικά πολύ λιγότερο από ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε στον χώρο αυτό. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, ενώ πριν από 10 χρόνια ήταν διαφορετική η κατάσταση. Υπήρχαν κενά 5 έως 6 ετών, τώρα όμως μιλάμε για δεκαετίες. Έχουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπω ότι εάν δεν στηρίξουμε τώρα την έρευνα στην ασφάλεια και την άμυνα και αν δεν διασφαλίσουμε κονδύλια γι' αυτό, τότε στο μέλλον θα απευθυνόμαστε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα ε, είναι αρεστό. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Ηνωμένε Πολιτείε θα είναι σε θέση να αφιερώσουν χρόνο και χρήμα για να προστατεύουν την Ευρώπη. Οι δικές μου ερωτήσεις τώρα. Μας είπατε ότι λείπουν πόροι. Ποιε λοιπόν θα ήταν οι προτεραιότητες στον χώρο της ασφάλειας και της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο θα καθορίσει αυτέ τις προτεραιότητες. Υπάρχουν πιέσεις από τον χώρο της βιομηχανίας, από διάφορα ε, ερευνητικά ιδρύματα, όμως δεν αντιστοιχούν απόλυτα στις ανάγκες στην άμυνα. Ποιος λοιπόν θα είναι αυτός που θα καθορίσει τις προτεραιότητες. Και έπειτα, μόλις αυτές οι προτεραιότητες γίνουν σαφείς. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή τη διαλογή όλων των προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ερευνητικά ιδρύματα, από την ε, βιομηχανία. Ποιος δηλαδή θα αποφασίσει για το ποιο έργο θα κερδίσει και θα αναπτυχθεί. Ένα ερώτημα ακόμα που θέλω να θέσω εγώ και αφορά τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία και τις λύσεις που πρέπει να αναζητηθούν. Μια προπαρασκευαστική δράση βασίζεται από τεχνική έποψη σε κάποιου κανόνες. Ποιου κανόνες θα διαλέξετε και ο μόνο τόπος όπου έχουμε τη σωστή αυτή ισορροπία που πρέπει να εξασφαλίσουμε σε ό,τι αφορά το, τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων για θέματα ασφαλείας και την ε, ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των κρατών σε ό,τι αφορά προμήθεια στρατιωτικού υλικού και τα πνευματικά δικαιώματα του ε, αμυντικού τομέα. Ήδη έχουμε πετύχει μια συμβαστική λύση που βασιζόταν και σε μια νομική αντιμετώπιση. Πρώτο ερώτημα. Ποιοι είναι οι κανόνες λοιπόν για την προπαρασκευαστική δράση. Δεύτερον, πιστεύετε ότι τα δικαιώματα πνευματικού χαρακτήρα για τον αμυντικό τομέα θα είναι διαφορετικά από αυτά που ισχύουν για τον πιστρατιωτικό τομέα. Και τέλος, σε πρακτικό επίπεδο, αναρωτιόμουν. Εγώ σας διαφο... διαβεβαιώνω το Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτή τη χρηματοδοτική πρόταση για την προπαρασκευαστική δράση. Αλλά σε σχέση με αυτό που κάναμε πριν από 10 χρόνια για τον τομέα έρευνας στην ασφάλεια, κάναμε μια πρώτη ενέργεια, αλλά στη συνέχεια δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση αυτών των προσπαθειών. Τώρα λοιπόν είναι κάπως εξωτικό που λέμε τώρα κάνουμε μια προπαρασκευαστική δράση αλλά εσωτερικά προσπαθούμε να περάσουμε τη γραμμή υφ, ε, για να βρούμε κάποια χρήματα στον προϋπολογισμό. Σε ποιο βαθμό λοιπόν θα μπορέσουν να υπάρξουν οι χρηματοδοτήσεις αυτές και η πρότασή σας πόσο θα κοστίσει όταν έρθει και από πού θα έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ για τα στοιχεία που μου δώσατε. Όπως είπα στην εισαγωγική μου παρέμβαση, είναι ένα θέμα για το οποίο εργαζόμαστε και δεν έχω συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Θα εργαστούμε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για όλα αυτά τα στοιχεία. Για το πιλωτικό σχέδιο τώρα. Σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Φορέα, είπαμε να καθυστερήσουμε λίγο περισσότερο την προθεσμία για να μπορέσουμε να δείξουμε ενδιαφέρον οι διάφορες εταιρείες γιατί η προθεσμία που είχε θεσπιστεί ήταν κάπως ε, σύντομη. Οι επιχειρήσεις μα υπέδειξαν θέλουν πιο πολύ χρόνο για να προετοιμαστούν. Δώσαμε λοιπόν αυτό το πρόσθετο χρονικό ορίζοντα, ο οποίο όμω δεν θα επηρεάσει καθόλου τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυλιχθεί η διαδικασία αυτή. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι προβλεπόταν, αλλά θα κερδίσουμε σε επίπεδο διαφάνειας και θα κάνουμε το λεγόμενο learning by doing, δηλαδή μάθηση δια του πράτην και αυτό θα μας βοηθήσει. Για την πρόταση προϋπολογισμού. Κομισιόν και θα πρέπει να υποβάλει ο πρόταση στις επόμενες εβδομάδες. Ποιο θα είναι το αριθμητικό ποσό, δεν ξέρετε, κυκλοφορούν μόνο φήμες. Οι φήμες όμως είναι από τη φύση τους φήμες. Αλλά από τη δική μας πλευρά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εμείς ζητούμε να διατηρηθεί το μέγιστο ποσό. Αυτό που είπαν οι προσωπικότητες, αυτό που εντόπισαν ως απαραίτητο. Αλλά για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, αν θέλουμε να μας πάρουν σοβαρά από την βιομηχανία, από τα κρατημέλη, από τον κόσμο της άμυνας, αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι σοβαρός. Αν έρθουμε με ένα γελίο προπολογισμό, θα είμαστε γελοί και είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε για να έχουμε ένα μέγιστο προπολογισμό για το, ήδη για το 2016. Για την ε, συμβουλευτική ομάδα, προ το παρόν η κυρία Μπιενκόφσκα δεν έχει πάρει θέση για το θέμα αυτό. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Είχε πει η κυρία Μπιενκόφσκα ότι θα σκεφτεί για το θέμα αυτό, αλλά προ το παρόν δεν υπάρχει οριστική θέση το πρόγραμμα, η Επιτροπή Προγράμματος έχει ήδη συνεδριάσει και κάναμε 4-5 συνεδριάσεις σχεδιασμού για το 2016 που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε περισσότερο για το πρόγραμμα εργασίας μας. Η συμβουλευτική ομάδα τώρα θεωρούμε ότι πρέπει ο κατάλογος των μελών του να οριστικοποιηθεί <clears throat> συντόμως Το θέμα δεν είναι αν θα έχουμε ένα άτομο περισσότερο, ένα άτομο λιγότερο. Συνεχίζεται η συζήτηση. Αλλά πιστεύω ότι προς το τέλος του Μαΐου, τέλος Ιουνίου καλύτερα, θα έχουμε τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων και θα συγκαλέσουμε μια πρώτη συνεδρία των εμπειρο, εμπειρογνωμόνων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι αυτή η ομάδα, γιατί θα μας δώσει την ανάδραση από τη βιομηχανία. είναι στο μέσο όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη μαθητείας και απόκτηση γνώσεων για μας και επομένως βασιζόμαστε στην ανάδραση από την βιομηχανία. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο προτιμούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικές ακόμα εβδομάδες, αλλά είμαστε σίγουροι ότι έχει μια σύνθεση που εκπροσωπεί πλήρως όλα τα συμφέροντα του αμυντικού τομέα. για τα αντικείμενα που θα αντιμετωπίσει ε, το εγχείρημα αυτό και γιατί είμαστε σε επαφή με τα κάτι μέρη και όχι με τον αμυντικό οργανισμό και με τους δύο. Βέβαια ο αμυντικός φορέας Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια πυρογνωμοσύνη την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Θα ήταν εκπληκτικό να παραγνωρίσουμε την εμπειρία αυτή και θα ήταν φάουλ να μην το κάνουμε. Αλλά από την άλλη έχουμε τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν και αυτά να εκφράσουν από τη δική τους άποψη, τη δική τους θέση και όπως ξέρετε η θέση ορισμένων κρατών μελών δεν συνάδει απόλυτα με την θέση του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Φορέα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας να εκφράσει την απόψή του. Συγχρηματοδότηση με τα κρατη αμφιβάλλουμε, έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Είναι κάτι που μας απασχολεί και αναλογιζόμαστε γι' αυτό, αλλά η συγχρηματοδότηση με τα κράτη-μέλη μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύπλοκη όταν μπλεχτούν και τα δικαιώματα πνευματικού χαρακτήρα. Γιατί αν τα κράτη-μέλη δώσουν χρήματα θα πούν και εγώ θέλω ένα μερίδιο από τα πνευματικά δικαιώματα αυτό θα συμπλεγματοποιήσει ακόμα περισσότερο το σχέδιο αυτό. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε λοιπόν αποκλείσει τελείως, αλλά θα είναι πολύπλοκο για να τεθεί σε εφαρμογή. Και το ερώτημα είναι αν αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο προπαρασκευαστικής δράση ή μεταγενέστρα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε. S'agissant du différentiel. Τώρα, Όσον αφορά το πώς θα γίνει η κατανομή, γιατί διαφορά υπάρχει μάλλον μεταξύ του, των όσων διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ε, είναι πολύ σημαντική, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον αμερικανικό προπολογισμό αλλά θα πρέπει να διακρίνεται το Ευρωπαϊκό προϋπολογισμός για να φτιαχτεί από συνοχή, από συνέπεια. Βεβαίω και είναι ανοιχτός ανταγωνισμός, οπότε θα πρέπει να υπάρχει πρικοδότηση αρκετή για την ε, προεπαρασκευαστική δράση, αλλά κυρίως να υπάρχουν κεφάλαια μετά, μετά τη δράση. Ε, διοικητικά μιλάμε για τέλος του 2016, οπότε το 2020 δεν είναι το αύριο ακριβώς, αλλά είναι το μεθαύριο. Άρα θα πρέπει ταχαίω να αρχίσουν τον ε, προβληματισμό, να επεσκεργαζόμαστε κάποιες προτάσεις για το τι θα γίνει μετά το 2020. Να γίνουν κάποιε σοβαρές προτάσεις, οπότε θα πρέπει να δούμε πω αυτή η ομάδα των προσωπικότητων θα καταλήξει σε κάποιε προτάσει σε κάποια νούμερα τα οποία και πρέπει στη συνέχεια να μας οδηγήσουν τώρα για τις ε, προτεραιότητες στην ε, έρευνα και ιδίω για την προπαρασκευαστική δράση. Βεβαίω και ποντάρουμε για άλλη μια φορά στην υπηρεσία μας γιατί έχει την εμπειρογνωμοσύνη θα πρέπει να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη αλλά και η βιομηχανία. Γι' αυτό και έχουμε ε, αυτό το όργανο συνεννόησης και με τα κρατημέλη και με την βιομηχανία και έτσι να καταλάβουμε κάποιες προτεραιότητες. Ένα σημαντικό στοιχείο ιδίω για την προβαστική δράση είναι οι προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να είναι περιορισμένες σε αριθμό. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν προπολογισμό ο οποίος θα πρέπει να είναι οριοθετημένο για να είναι αποτελεσματικό για να είναι συνεπή. Επομένω θα πρέπει να περιοριστούμε σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα εκεί να επικεντρώσουμε και δημιουργικά τι προσπάθειε και να δούμε ε, πώ μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα θα έχουμε καλές επιδόσεις. Τώρα όσον αφορά για του κανόνε οι οποίε θα διέπουν τα, ε, τις ε, δημόσιες συμβάσεις, την πνευματική ιδιοκτησία κλπ. Το 2020 είναι κάτι βασικό, αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα της ρύθμισης που θα μας διέπει, γιατί τα συζητάμε τα κράτη-μέλη και την βιομηχανία για το πώς θα φτιάξουμε ένα σύστημα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας που θα ανταποκρίνεται τις ανάγκες αυτού του τομέα της άμυνας. Τα στοιχεία για τις λεπτομέρειες δεν τα έχουμε όλα, καλά κρατούν οι συζητήσεις, οπότε θα δοθεί ένα ε, σχήμα ε, σε αυτή την σύλληψη. Ε, μόλις αποφασίσει η Ευρωπαϊκή δεύτερο εξάμεινο. Αλλά θα πρόκειται να προσαρμόσουμε το τι θα ισχύσει στις ανάγκες της ε, άμυνας. Πάρα πολύ βασικό είναι ότι σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις για την άμυνα από πλευράς οικονομικής δεν είναι πραγματικά μια αγορά με ζήτηση και προσφορά. Στην αλήθεια πρόκειται για κάποια όσμωση, κάποια συνεργασία μεταξύ Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και της Βιομηχανίας. Οπότε και εμείς θα πρέπει την διάσταση πραγματικότητα να την πάρουμε υπόψη, μια που κατά 90% οι παραγγελίες του, του κλάδου και της βιομηχανίας εξαρτώνται και δίνονται από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας. Ο Πρόεδρος. Μάλιστα, δεν ήσασταν αρκετά ακριβή στην απάντησή σας για τη συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία, ε, Εάν αυτή τη στιγμή διατεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για προπαρασκευαστικές δράσεις, θα πρέπει να υπόκειται σε κάποιον ε, δημοσιονομικό κανονισμό, είτε δηλαδή ε, τον προπολογισμό είτε κάποιες παρεκκλήσει. Για, τα, τα PPPs, για παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σα ερωτώ απλά ποιοι είναι οι κανόνε συμμετοχής Στου οποίους θα βασιστούν αυτές οι προπαρασκευαστικές δράσεις και τη χρηματοδότησή τους και στα πλαίσια αυτών των ε, δράσεων. Δεν γίνεται να διαπραγματευτούμε με τα κράτη-μέλη, διότι θα βασίζεται η χρηματοδότηση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος δεν επαναδιαπραγματεύεται. Άρα λοιπόν, ο γενικός προϋπολογισμός είναι εκεί που θα στηριχτεί αυτή η προπασκευτική δράση ή κάτι άλλο, ή θα ζητήσετε μια παρέκκληση, μια εξαίρεση από τα, που πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη και από το Κοινοβούλιο. Και παρομοίως με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. εάν προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρχουν, θα διέπεται από κάποιους κανόνες και πρέπει να βρεθεί λύση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ρωτώ ποιοι είναι οι κανόνες στους οποίους θα βασίζεται ε, η χρηματοδότηση. Πώς θα δίδονται τα κονδύλια, διότι διαφορετικά ε, χανόμαστε. Μας είπατε κι εσείς ότι η αγορά δεν είναι τέλεια, ότι υπάρχουν προβλήματα, όμως ο προϋπολογισμός και οι ε, κανόνες που τον διέπουν σχετικά με τη χρηματοδότηση δεν έχουν αλλάξει. Υπάρχει κάποια σκέψη ανάμεσα στα κράτη-μέλη σχετικά με τις ε, λεπτομέρειες, ε, σχετικά με το από πού θα έρθει η χρηματοδότηση, θα γίνεται κάποιος διαγωνισμός. Στα πλαίσια όμως του ευρωπαϊκού προπολογισμού δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια ευελιξία. Υπάρχει προπολογισμό ο οποίο ε, καταρτίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Ποιοι είναι οι κανόνε λοιπόν στους οποίους θα βασιστεί η χρηματοδότηση για τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Ο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, πούμε, θα μπορούσε να δει, να αποβάλει κάποια πρόταση για το πώ θα βρεθεί η χρηματοδότηση. Ε, ο κύριος Γκάλερ. Ναι, σύντομα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Μας είπατε ότι ο προπολογισμό αυτός ε, θα ε, είναι κάτι με το οποίο θα το 2017 2017-2018 και έπειτα. Υπάρχουν όμως κάποια κενά μέχρι τότε. Θα βασιστεί δηλαδή ε, η χρηματοδότηση στο άρθρο 185 προβλέπει χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο κύριος Αλέξης. Για τη συγκεκριμένη νομική βάση, αυτό είναι το τμήμα των θεμάτων που παραμένουν ανοιχτά. Συνεργαζόμαστε ακόμα για τα θέματα αυτά και θα πρέπει σε επόμενες εβδομάδες να καταλήξουμε σε μια θέση για το θέμα αυτό. Αν με ξανακαλέσετε σε λίγε εβδομάδες, κάτι θα έχω να σας πω πάλι. Πιο συγκεκριμένο. Για την περίοδο χάσματος. Αυτά που είπατε είναι μία δυνατή οδός. Αλλά δεν έχουμε ακόμα περατώσει τα θέματα στα οποία έχει ολοκληρωθεί η σκέψη μας για το 2017 και την ε, ε, προπαρασκευαστική δράση. Είναι ένα χένον χάσμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα που θέλετε να θέσετε. Κάποια πρόταση, κάποια δήλωση. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, as a compliment... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Αλέξης Μπορώ να σας ε, επιβεβαιώσω ότι έχει γίνει πρόοδο σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητε του, προγραμμα... του προγράμματος. Ο στόχος μα είναι να έχουμε διάλογο και, και brainstorming με τα κράτη-μέλη. Πρέπει να δούμε ποια είναι η σύνδεση με τη δημιουργία ικανοτήτων και την ΚΕΠΑ, ώστε θα οργανώνουμε μηνιαίες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων, εμπειρογνωμόνων από τη βιομηχανία, τα Υπουργεία Άμυνας, για να δούμε αν υπάρχει κάποια σύγκληση στα θέματα αυτά και οι πληροφορίες αυτές διαδίδονται στην Κομισιόν για να τις εξετάσει. Τρεις συναντήσεις είχαμε μέχρι στιγμής, Μάρτιο, Απρίλιο και μία ένα εργαστήριο δύο ημερών το Μάιο και ρωτήσατε πώς σκεφτόμαστε για την εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό θα ακολουθήσει τις συμφωνίες των εθνικών αντιπροσωπιών, μάλλον τις ε, συμφωνίες για εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια συμφωνία που καθορίζει τι θα κάνουμε. Έχουμε εξετάσει εναλλακτικέ λύσεις για το πρόγραμμα εργασίας και μετά η αρμόδια επιτροπή θα διαλέξει τα θέματα τα οποία θα είναι το αντικείμενο, θα ακολουθήσει και μια πρόσκληση ενδιαφέροντος και μια φάση αξιολόγησης. Το θα κάνω λοιπόν και για την προπαρασκευαστική δράση, όταν είναι έτοιμες οι συμφωνίες αυτές για την εκκόρυψη θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή των ενεργειών. Είμαστε έτοιμοι και η μονάδα μας ασχολείται με το θέμα αυτό και προσπαθούμε να προκαταλάβουμε αυτά τα οποία θα λάβουν χώρα. Να προσθέσω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον αμυντικό φορέα να έχει ένα σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα. Θέλουμε να αναφερθούμε και στην έκθεση GAP και στο, στη διάσκεψη κορυφής Γαλλίας-Γερμανίας που ζήτησε ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Έχω και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή να οθήσουμε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση στον ορίζοντα 2020 για παράδειγμα υπάρχουν αυτά τα PPP, προβλέπετε να παίρνει κάποιος κάποια παρέκκληση από τους κανόνες. Τι θα γίνει, θα υπάρχει συνεργασία με ένα περιορισμένο αριθμό κρατών μελών που θα συνεργάζονται υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ε, υπό το άρθρο 184, ας πούμε που αναφέρεται στο πρόγραμμα πλαίσιο. Και το άρθρο αυτό επίσης προβλέπει τη δυνατότητα μιας ε, ομάδας με περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, η οποία θα εργάζεται έτσι. Εξετάζεται και αυτά τα ενδεχόμενα. Αλέξης. Οπωσδήποτε αυτό είναι βάση για προβληματισμό. Πρέπει επομένως όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη και για την ε, ε, προπαρασκευαστική δράση αλλά ίσως και για την περίοδο μετά την προπαρασκευαστική δράση. Οπότε και η επιτυχία της δράσης βεβαίως και εξαρτάται από το πόσο απλή είναι. Η πρικοδοτή θα είναι τόσο τρομερή σε σχέση με τις ανάγκες του κλάδου. Άρα μάλλον θα πρέπει να περιορίσουμε τις ε, περιπτώσεις και πιθανότητες ε, παρέμβασης. Τέλος πάντων η ιδέα υπάρχει, την κρατάμε, θα είμαστε προσεκτικοί. Ο Πρόεδρος. Ωραία. Όλοι μας είμαστε επιφυλακτικοί μένα αλλά έχουμε ενδιαφερθεί πάρα πολύ από αυτά που είπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους αυτούς που σε μία δύσκολη Δευτέρα απόγευμα ήρθατε εδώ να ακούσουμε και τον κύριο Αλέξη και το Κοινοβούλιο φυσικά περιμένει σε επικείμενες προτάσεις που θα έρθουν από την Κομισιόν και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της νομοθετικής περίοδου το νωρίτερο ίσως πριν από το τέλος της ε, πριν από το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε αυτή την πρόταση από την Κομισιόν. Υπάρχει κάποια άλλη αίτηση, πρόταση, σύσταση. Εντάξει, σας ευχαριστώ λοιπόν για την συμμετοχή σας και θα τα πούμε στις 15 Ιουνίου, 9 η ώρα το πρωί. Τσίς.